Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής έχουν καταφτάσει, οπότε κηρύσω την έναρξή της. Θα ήθελα να επενθυμίσω το αντικείμενό της. Πρόκειται για το συγκρότηση σε σώμα του Προεδρείου της Επιτροπής, της Δικής Επιτροπής για τις εκπομπές των οχημάτων, φυσικά με εκλογή Προέδρων και Αντιπροέδρου, Προέδρου και Αντιπροέδρων, βάσει των άρθρων 198 και 204 του ιστορικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ακολουθήσουμε φυσικά τη σειρά πρώτα, ε, πρόεδρος και στη συνέχεια αντιπρόεδρε. Οι πολιτικές ομάδες ε, έχουν ορίσει κάποια μέλη, όπως ο κύριος Βιν Βαντεκάβα που ε, αντικαθίσταται από την κυρία Κλούν, η κυρία Μοντέρο Ντεαγκιάρ που αντικαθίσταται από τον κύριο Γκάμπους για το ΕΛΚ αυτά στους σοσιαλιστέ και δημοκράτες Μάσιμο Παολούτσι ε, που αντικαθίσταται από τον Νίκολα Ντάντι και από το ΙΕΝΕΦ Γιώργ Μαγέρ που αντικαθίσταται από τον Μάριο Μπουργέζιο. Βλέπω ότι γνέφεται όλοι καταφατικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να εξακριβώσω πρώτα απ' όλα ότι έχετε τις κάρτες σας μαζί για την ψηφοφορία, διότι θα τις χρειαστούμε. Πολύ ωραία. Θα πρέπει να εξακριβώσουμε την απαρτία 12 άτομα, κανένα πρόβλημα, είναι πολύ πιο αδρό η προσέλευση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε τώρα τις υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Ποιος είναι υποψήφιος. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να ορίσω την Κάθλιν Φαν Πρέμπτ στη θέση υποψηφίου για την Προεδρία της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Ο κύριος Κάρινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στο βάση του της γενικής συνεργασίας που επικρατεί στο Κοινοβούλιο το ΕΛΚΑ δεν αντιτάσσεται στο διορισμό της κυρίας Κάθλιν Βαν Πρέντ στη θέση της υποψηφίου για την Προεδρία της Επιτροπής. Παρόλα αυτά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι το ΕΛΚΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να μην επιτρέψει το κυνήγι των μαγισσών μέσα σε αυτή την Επιτροπή κατά της βιομηχανίας ή κατά της τεχνολογίας του ντίζελ όπου έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εδώ στην Ευρώπη σε παγκόσμια κλίμακα γιατί θα ήταν λάθος να έχουμε αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στη βιομηχανία και στο περιβάλλον. Ο, το καθήκον μας ε, είναι να, ε, υπάρχει, να συμβαδίζει η βιομηχανία με τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Οι σοσιαλιστές έχουν υποβάλει λοιπόν επίσημα την υποψηφιότητα της Κάθλιν Βαν Μπρέντ. Συμφωνείτε κυρία Βαν Μπρέντ. Βεβαίως ε, πρόεδρε. Συμφωνώ. Διαπίστωσα λοιπόν πως ε, η υποψήφια έχει υποβάλει και την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τυπικό. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε τώρα στην εκλογή του της Προέδρου της Επιτροπής, διότι έχουμε μία, μία μόνο υποψήφια. Για λοιπόν θα εκλέξουμε την Πρόεδρο της Επιτροπής. Donc personne n'ayant réclamé le vote à bulletin secret, euh, eh bien... Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, κυρία Φαν Μπρέντ για την ε, εκλογή της, ταχύτατη αυτή εκλογή. Παρακαλώ, ελάτε στο Προεδρείο, εμένα έληξε ο ρόλος μου. Good morning, uh, dear colleagues. Um, not... Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρόκειται να εκφωνήσω λόγο μεν. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου όμως για, τις, ε, για την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων δε. Ιδιαίτερα στρέφουμε και προς το ΕΛΚ και προς τους ε, συναδέλφους αυτής της πολύ σημαντικής ερευνητικής επιτροπής. Σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι πρόεδρος της διαφάνειας, της, ε, ε του ανοίγματο, θα συνεργαστώ με τον κάθε έναν και την κάθε μία εδώ και στο Προεδρείο και στην Επιτροπή να γίνει μια ουσιαστική ερευνητική επιτροπή, συμφωνούμε απολύτως. Θέλουμε να δουλέψει λοιπόν αυτή η επιτροπή κατά τρόπο αποτελεσματικό και να επιτύχει αυτά που θέλουμε να επιτύχει ώστε στο μέλλον να έχουμε καλύτερη υλοποίηση και εφαρμογή και επιβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και σας ευχαριστώ. Ας περάσουμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροέδρων, όπως υπόθηκε και νωρίτερα. Απαρτία έχουμε. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με τους αναπληρωτές. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε Ποιος είναι υποψήφιος για τη θέση του πρώτου... Ε, με συγχωρείτε που κάνω και λαφάκια, δεν είμαι συνηθισμένη. Για τη θέση του πρώτου του Πρόεδρου, κύριε Κάριν. Πρόεδρε, ευχαριστώ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Ιβο Μπέλετ. Very much. Mr. Bellet. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέλετ. Δέχεστε αυτή την υποψηφιότητα. Μάλιστα λέει ο κύριος Μπέλετ. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι από άλλες πολιτικές ομάδες. Όχι. Μπορούμε λοιπόν διαβοής να επιβεβαιώσουμε την εκλογή αυτή. Ήβο, σε παρακαλώ να έρθεις εδώ, κοντά μου. it will only get worse. well, it's Flemish, but. Um, Okay, then I can go to the election of the second. Περνώ λοιπόν στην εκλογή δεύτερου αντιπρόεδρου. Έχετε υποψήφιο. Παρακαλώ κύριε Χένκελ. Εκ μέρους ομάδας των συντηρητικών μεταρρυθμιστών θέλω να προτείνω τον κύριο Ντεμέσμέκερ. Πάλι Ολλανδικά. Do you agree? Συμφωνείτε κύριε Ντεμεσμέκερ. Ναι βεβαίως βεβαίως και συμφωνώ. Φαντάστες. Um, are there any other candidates from other political... Πολύ ωραία και υπάρχουν άλλοι υποψήφοι από άλλη πολιτική ομάδα. Όχι. Η Επιτροπή δέχεται διαβοή στην εκλογή, ναι, και παρακαλώ Μάρκ, έλα. No, the Flemish Parliament. But this is not the natural coalition of the Flemish Parliament. In the future. In the future. Can I now move for the election? Τώρα μπορούμε να περάσουμε στην εκλογή τρίτου αντιπρόεδρου. Υπάρχει υποψήφιο. Dear Chair, dear colleagues, uh, Πρόεδρε, η Γκουε προτείνει την Κατερίνα Κονέτσινα. Ε, για να αλλάζουμε και φίλο και γλώσσα, παρεμπιπτόντως. Ναι, δυστυχώς δεν γνωρίζω τη γλώσσα σας, αλλά θα πρέπει να τη ρωτήσω εάν συμφωνεί. Καλός έτερος υποψήφιο υπάρχει. Όχι, λοιπόν, διαβοής παρακαλώ. And please join us. Um... Και περάστε. absolutely. Okay, can I go for the election of the last and the fourth? Τέταρτος και τελευταίος αντιπρόεδρος. Κύριε Χάουτ, τι έχετε να πείτε. Ω, καλημέρα σας και καλημέρα σας. Χαίρομαι που ακούω τόσα φλαμανδικά στο Προεδρείο. Και γι' αυτό προτείνω άλλη γλώσσα. Εμείς ως πράσινοι προτείνουμε την ε, Κάρι Μαντελή ως τέταρτη αντιπρόεδρο στα γαλλικά. Κύριε Αντελή, δέχεστε την υποψηφιότητα αυτή. Ναι, ναι, τη δέχομαι. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, αφού δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, ας εγκρίνουμε και αυτή την υποψηφιότητα διαβοής και σας ευχαριστώ. Well, colleagues, um, amazingly smooth, um, and thank you very much. Oh, of course you should. Και παρακαλώ να έρθετε και εσείς κοντά μας. Βιάζομαι, βιάζομαι. Dear colleagues, um, the only thing that um, keeps us... Συνάδελφοι, το μόνο που μας κρατάει μακριά από ένα καφεδάκι είναι οι ανακοινώσει. Θέλω να σας πω ότι η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής θα γίνει την 3η 22 Μαρτίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Οι συντονιστές και το Προεδρείο θα προτείνουν ε, το ατζέντα μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα σας έχουμε ετοιμάσει πρόταση μέχρι τότε, αλλά έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας γιατί πρέπει να συστήσουμε τη μεθοδολογία, να αποφασίσουμε πώς θα δουλέψουμε, ποιον θα καλέσουμε ε, και βέβαια όλα αυτά ήδη τρέχουν, αλλά η πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει είναι η συνεδρίαση των συντονιστών και αυτή θα γίνει στο Στρασβούργο την επόμενη Πέμπτη στις 10 Μαρτίου από τις 10 μέχρι πριν τις ψηφοφορίες, λίγο πριν τις 12 δηλαδή. Και φυσικά είστε όλοι ε, προσκεκλημένοι. Θα σας ενημερώσει η γραμματεία για το πού και πότε. Μπορείτε ήδη να το σημειώσετε όμως στην ημερήσια σας, ε, στο πρόγραμμά σας. Η ατζέντα θα είναι η πρώτη συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή σε αυτήν την Ερευνητική Επιτροπή. Θα έχουμε ένα σύνολο προτάσεων που θα είναι έτοιμο μέχρι τότε. Βέβαια για να μπορέσουμε να συγκαλέσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών είναι σημαντικό κάθε πολιτική ομάδα να μας ανακοινώσει ποιος θα είναι ο συντονιστής της, ε, στη Γραμματεία και στο ε, Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στις 22 Μαρτίου.